Επίτροπε, συνεχίζουμε την συνεδρίασή μας. Τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης και τα κείμενα που έχουν εγκριθεί είναι διαθέσιμα. Δεν βλέπω κάποιος να θέλει να κάνει σχόλια σχετικά. Επομένως εγκρίνονται τα χθεσινά πρακτικά.